Good afternoon, colleagues. Can I call the meeting to order? First and foremost, Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε, είναι το σημαντικότερο, πρώτο σημείο, για την έγκριση της μερικής διάταξης. Συμφωνείτε, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο. έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 10 και 11 Οκτωβρίου. Εγκρίνονται. Σας ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Λευκή βίβλος για το μέλλον ε, της πολιτικής μεταφορών. Ο κύριος Γκρός ε, για να συζητήσουν στροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με βοήθησαν ως και οδησηγητές και οι οποίοι έδειξαν και τώρα πνεύμα συνεργασία στην αναζήτηση των τροπολογιών και των συμβασμών στις τροπολογίες. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστώ και το δικό μου προσωπικό αλλά και τη γραμματεία που έκαναν πολύ καλή δουλειά έτσι ώστε οι 413 τροπολογίες να περιοριστούν σε 32 συμβαστικές. οι οποίες καλύπτουν 288 τροπολογίες. Αυτές οι 32 συμβαστικές. Πολύ καλή δουλειά λοιπόν. Και ελπίζω ότι θα έχουμε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα μια ναι, σύντομη δηλαδή γνωμοδότηση όπως ελπίζουμε για τη Λευκή Βίβλο, 40 σελίδες το πολύ, με τις πολιτικές, τα πολιτικά χαρακτηριστικά που διεκδικούμε. Δεν θα επισέλθω στις ε, λεπτομέρειες στο περιεχόμενο. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι ίσως κάποιοι να ε, θεωρήσουν ότι δεν καλύπτονται απόλυτα από μια συμβαστική τροπολογία γιατί δεν αντικατοπτρίζει τη δική τους τροπολογία. Θα το δούμε στην ψηφοφορία αυτό, αλλά πάντως ελπίζω να είναι ικανοποιημένοι περισσότεροι και θα δούμε και για την ψηφοφορία αύριο περίπου, αύριο το πολύ θα έχουμε έτοιμη και την, ε, έτοιμες και τις προστάσεις μας. Για τις υπηρεσίες λοιπόν, λιμένων. Ξέρετε ότι πολλοί συνάδελφοι δεν συμφωνούν με την απελευθέρωση με αυτού. Άλλοι θεωρούν ότι αυτά τα οποία έχει περιλάβει σε προηγούμενο έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αναπτυχθούν σε περισσότερα έγγραφα, τρία-τέσσερα έγγραφα από την Επιτροπή. Άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να αφήσουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει συνένεση και μάλιστα και μέσα σε ορισμένες πολιτικές ομάδες ε, παρουσιάζονται αποκλίνουσε απόψει. απόψεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πριν να ε, προσέλθει με την νομοθετική της πρόταση σε δύο χρόνια περίπου όπως είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ λοιπόν προτείνω το 2012 να φροντίσει να μας ενημερώσει για τις προθέσεις της μέσα στο επόμενο έτος, έτσι ώστε να δούμε τι σκοπεύει να πράξει προς το θέμα της απελευθερώσεων των λιμενικών υπηρεσιών για να έχουμε περισσότερο χρόνο στη θέση μας να, τη συζητήσουμε. Επίσης από πολλούς οικονομικούς κύκλους ακούγεται ενδιαφέρον για αυτή την εκδήλωση προθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως είπα, όχι σε λεπτομέρειες, αλλά να ξέρουμε τι μπορεί να μας περιμένει από εδώ και μπρος. Και θα ήταν καλό να ακούσουμε και αυτούς τους οικονομικούς κύκλους και τις θέσεις τους ως προς την πρόταση της Επιτροπής. και δεν με ενδιαφέρει να επιλέξω την απελευθέρωση ή τη μία απελευθέρωση δομέα των λιμενικών υπηρεσιών, αλλά πάνω απ' όλα να μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αυτό είναι για την 26, για την 33, υπαριθμόν τροπολογία, ε, 23, ε, για το πολυλειτουργικό σύστημα. Θα ήταν καλό να είμαστε πιο συγκεκριμένοι μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Γιατί ορισμένα πράγματα θα εξαρτηθούν πιστεύω και από την Επιτροπή και πάντως είναι αρκετά σημαντικό το θέμα. Για την, ε, για την τροπολογία 24, όσον αφορά την διαμετακόμιση και την απελευθέρωση της μετακόμισης, θα ήταν καλό να επανέλθουμε και να δούμε αυτά τα οποία είχαμε πει στην Επιτροπή μας και στις προφορίες μας, ότι θα πρέπει δηλαδή η διαμετακόμιση να απελευθερωθεί όταν έχουν επιληθεί και τα λοιπά ζητήματα που συνδέονται, κοινωνικά προβλήματα κτλ. Το καποτάζ δηλαδή. Γιατί είναι πολλές οι διαστάσεις του ζητήματος. Και πιστεύω ότι η συζήτηση με τον προκάτοχό μου τότε και τον πρόεδρο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, για το πώς λέει, θα μπορούσαμε να έχουμε καλούς κανόνες, καλές διατάξεις, εναρμονισμένες διατάξεις στο με αυτό. Υπ' αυτέ τι συνθήκε λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα έτσι ώστε και να τηρήσουμε τόσο έχουμε συζητήσει και να είμαστε σαφείς. Για τις πολυλειτουργικές μεταφορές ε, δεν ισχύει το ότι διαφωνούσαμε τα 300 χιλιόμετρα όπως, ε, όπως ε, είχε ακουστεί. Αλλά να έχουμε μία κατανομή ε, διαλειτουργική, ικανοποιητική στις μεταφορές. Και σε αυτό πιστεύω ότι έχουμε ευρύτερη υποστήριξη και στη συμβαστική τροπολογία για το θέμα αυτό. Στην επόμενη συμβαστική, στη 10 δηλαδή, Connecting Europe Facilities, θα ήθελα να επισημάνω ότι Και σε αυτό θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια ικανοποιητική συμβαστική, αλλά και για τα project bonds και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον αναφέρεται στα project bonds και όχι στα euro bonds, όχι στα ευρωομόλογα δηλαδή, αλλά στα ομόλογα που αφορούν ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό ε, σχέδιο ή πρόγραμμα. Αυτά τα project bonds ε, υποστηρίζουμε εμείς και όχι τα ευρωομόλογα. Αυτά είναι τα κύρια σημεία. Έχετε δει τον κατάλογο των, τροπο, των ψηφοφοριών και εσείς και πιστεύω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ευρύτερη πλειοψηφία στο θέμα αυτό. Σημαντικό επίση θα ήταν να υπογραμμίσω ότι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο πρωί δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουν, να επαραληφθούν. Αυτά τα οποία είναι σημαντικά τα υπογραμμίζουμε επαρκώ. Και Εν τέλει, σημειώνουμε ότι αναμένουμε μία πρόταση από την Επιτροπή και άρα δεν προχωρούμε σε ανάπτυξη των θέσεών μας ως προς το τι θα πρέπει να είναι αυτή η πρόταση της Επιτροπής. Μια θέση λοιπόν ρεαλιστική. Ξέρω βέβαια ότι η Επιτροπή τα βλέπει κάπως πιο στενά όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει ένα άλλο θέμα, μια ερώτηση περισσότερο συναδέλφου τη σημερινή συνάντηση των συντονιστών από το ΕΛΚ ε, και όχι τροπολογία. Στα δύο δηλαδή σημεία στα οποία ανεβλήθη η συζήτηση και δεν θα ήθελα να ξαναρχίσω όλη τη συζήτηση βέβαια την ε, αποδεσμοποίηση αλλά και την ε, ανάπτυξη των αγορών στην οποία έχουμε αναφερθεί, ως προς την αποδεσμοποίηση που πάλι υποτίθεται ότι θα μας καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 και μετά μία ε, τροπολογία, δεν καλύπτει το θέμα της ε, απελευθέρωσης των αγορών. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι οι συνάδελφοι του ΕΛΚ ενδιαφέρονται να δούνε πού τίνει η υπόθεση χωρίς να λαμβάνουμε θέση ε, για το θέμα αυτό συγκεκριμένο. Αυτά και ελπίζω να ακούσω και τις δικές σας θέσεις και πάλι ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία στον, στην επεξεργασία των συμβαστικών τροπολογιών. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκρός ο Αλκαντράουι από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω καταρχάς ε, συγγνώμη εκ μέρους ε, της συναδέλφου Σανελόπρου, η οποία δεν είναι εδώ. Αλλά εγώ εκ μέρους της δικής μου πολιτικής ομάδας θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει και γιατί έδειξε προθυμία να συνεργαστεί μαζί μας αλλά και με τις άλλες πολιτικές ομάδες ώστε να καταλήξουμε σε καλές συμβιβαστικέ προτάσεις. Εξακολουθούμε, μάλλον μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ε, εξακολουθούσαμε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας και χαίρομαι και είναι πολύ επικοδομητική η στάση της, γιατί τις περιέλαβε και τις τελευταίες μας προτάσεις στην εξέταση των τροπολογιών. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, έχω να κάνω μια πρόταση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να εγκριθεί η διατύπωση στην παράγραφο ε, που δεν θα λέει για απελευθέρωση, αλλά ότι θα λαμβάνονται υπόψη καθολικέ υπηρεσίε κτλ. Τέλο πάντων, να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση που έχουμε χρησιμοποιήσει και κατά το παρελθόν για να αποφύγουμε προβλήματα με τη διατύπωση. Τώρα, κάποια σχόλια σε σχέση με κάποιε άλλε συμβαστικέ προτάσει συμφωνούμε με αυτό που είπατε για το κατόφλι των 300 χιλιόμετρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνει μια καλή πρόταση ευρυατενία διότι θέλει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για τους σιδηροδρόμους στις μακρές αποστάσεις αλλά για τις ε, βραχύτερες αποστάσεις μπορεί να σημειωθεί μεγάλη πρόοδος πιστεύω και εντός των κρατών μελών άρα συμφωνώ πλήρως με τη δική σας πρόταση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα, πολύ, ε, τα giga liners, ε, τα πολύ μεγάλα αυτά πλοία, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Και δεν νομίζω θα υποστηρίξουμε την ιδέα αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα την συμβαστική υπαριθμών 22, Λέτε ότι κάποιες αλλαγές ε, σε σχέση με τις διαστάσεις των οχημάτων. Θα πρέπει να βοηθήσουν ώστε και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα. Αυτό είναι σημαντικό και να μειωθούν εκπομπές. Αλλά σε ό,τι αφορά την 23 δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Δεν θα προκληθεί και καμία επανάσταση βέβαια από αυτό, απλά εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα ως ομάδα. Δεν είμαστε υπέρ αυτών των gigaliners. Σε ό,τι αφορά τώρα τις λιμενικές υπηρεσίες, γνωρίζετε ότι η ομάδα μου δεν διακατέχτηκε από ιδιαίτερο ενθουσιασμό για μια επανέναρξη συζήτηση σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Βέβαια, εναπόκειται στην Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσο θέλει να προχωρήσει σε περαιτέρω συζήτηση, να αναθέσει ίσω τη διεξαγωγή περαιτέρω μελετών, να η συζήτηση διαπραγματεύσει με του εμπλεκομένου φορεί. Εμεί πάντω δεν θα θέλαμε να τεθεί συγκεκριμένο αίτημα στην Επιτροπή για να, αντιμετωπι... για να εξετάσει αυτό το θέμα. Χαιρόμαστε που συμπερίληθησαν ε, τα ομόλογα έργων. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Σε ό,τι αφορά τα συμβιβαστική 18 για τα δικαιώματα των επιβατών, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τις ενέργειες μεταφορές, ίσως το μέλλον και σε άλλες μορφές μεταφορών, Υπάρχει ένα επιπλέον κόστος το οποίο μετακυλείται στον επιβάτη. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα στηρίζουμε 100% τη μικρή αυτή αλλαγή στο κείμενο. Σε ό,τι αφορά τη συμβιβαστική 24 για τις οδικές μεταφορές, υποστηρίζουμε την τελευταία εκδοχή που αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο. Ε, για τις ώρες ε, οδηγήσεως και αναπαύσεως, να αλλάξει δηλαδή το πλαίσιο. Και σε ό,τι αφορά την, ε, το πλαίσιο αυτό λοιπόν, είδαμε την περσινή έρευνα που έγινε και που έδειξε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις ό,τι αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και την εφαρμογή των κανονισμών. Δεν υπάρχει δηλαδή εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν εξετάσουμε τις εργασιακές συνθήκες ε, θα πρέπει να βελτιωθούν βέβαια και τα κοινωνικά, ε, οι κοινωνικέ πτυχέ ε, για του εργαζομένου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να κάνω. Συνολικά πρέπει να πω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά με τον εισηγητή. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο γι' αυτό και πιστεύω ότι η έκθεση θα εκπέμψει ένα πολύ καλό μήνυμα από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου για το τι θέλουμε ε, να επεξεργαστεί ακόμη περισσότερο η Κομισιόν και που θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Ευχαριστώ. Κυρία Μάισνερ από την ομάδα Άλντε τώρα. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ θερμά εκ μέρους ομάδας με τον Ματσίου. Είναι πάρα πολύ ικανός, όχι μόνο ως προς την πολιτική, αλλά και ως προς τη διπλωματική πτυχή του ζητήματος. Είχαμε πολλές προτάσεις από διαφορετικές ομάδες. Άλλοι ήθελαν περισσότερη έμφαση στο περιβάλλον, άλλοι στο, στα κοινωνικά, άλλοι περισσότερη απελευθέρωση. Διαφορετικέ τάσει, οι οποίε αντιστοιχούν τελευταίο και με τι πολιτικέ θέσει των πολιτικών ομάδων. Αλλά κατάφερε ο συνάδελφο Γκρό να τα χειριστεί όλα με πολύ μεγάλη επιδεξιότητα και να καταλήξει σε ικανοποιητικέ συμβαστικέ τροπολογίε. Δεν θα αναφερθώ στα όσα είπε διεξοδικά και ο κύριο Γκρό και ο κύριο Ελκαντράουι. Απλώ ένα-δύο σημεία όπου θεωρώ Φερρυπίν καλό το ότι ε, τώρα αναφέρονται τα 300 χιλιόμετρα, δηλαδή λέμε στη συμβαστική τροπολογία ότι μπορεί κανείς να έχει ε, πιο σύντομες και οικολογικές λύσεις ή εναλλακτικέ. Για τα μεγάλα φορτηγά, για τα πολύ μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα πάλι είναι σαφές για μας ότι θέλουμε και να τα χρησιμοποιούμε βεβαίω για να υπάρχει εξοικονόμηση ενέργεια, αλλά μόνο σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Δεν πρέπει δηλαδή η ζωή μα να γίνει και πιο επικίνδυνη από τη χρήση του. Αυτό είναι καλή συμβαστική δηλαδή που βρέθηκε. Και επίση ένα-δύο πράγματα ακόμα συγκεκριμένα. 153 σελίδα, σελίδα 8 συγκεκριμένα τη κυρία Γκρίσπατ. Ε, έχω βλέπω ένα πρόβλημα μετάφραση εδώ. Γιατί ε, αντιπαραθέσαμε το γαλλικό που το αυθεντικό κείμενο και το αγγλικό. Στο αγγλικό λέει could, θα μπορούσε. Μπορεί. Αλλά νομίζω ότι με βάση την αρχή του use it or lose it, δηλαδή πει την ευκαιρία ή χάνεται, ε, θα έπρεπε να είμαστε πιο αυστηροί. Όπως είναι το γαλλικό κείμενο. Συμφωνεί λοιπόν ο εισηγητής να το ε, προσαρμόσουμε. Λυπάμαι που υπαρξήφισε αυτό το λάθος, αλλά θα μπορούσαμε νομίζω να το δούμε. Στη σελίδα 10 του κυρίου Τρεμόσα. Μήπως έχει αποσυρθεί. Δεν είναι εδώ ίδιος για να μας πει το 199, η 199 τροπολογία να έχει αποσυρθεί, αλλά φαντάζομαι θα μας ενημερώσει. Σελίδα 11. Ναι, ε, αναφέρομαι στους καταλόγους των ψηφοφοριών. σελίδε 8 και 10 του καταλόγου ψηφοφοριών που δεν έχουν διερμηνεί. Και προχωρώ στην 11. Στην 24 τη κυρία Γκρίσπακ πάλι υπάρχει κάποια παρερμηνία. Γιατί ξέρω ότι ήθελε να διαγράψει αναφέρεται όμως, ε, ήθελα να διαγράψει το, την αναφορά στην Ευρώπη ως κέντρου καινοτομίας κτλ. Ενώ ε, βλέπουμε τώρα στο 266 ότι ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα από αυτό που επεδίωκε οι ενδιαφερόμενοι. Ίσως θα πρέπει να διευθυνθεί αυτό. Στην δε συνέχεια είχαμε συμφωνήσει στην 26Β μια σημαντική τροπολογία που θα ψηφιζόταν σε τμήματα. Ξέρω ότι δεν είναι εδώ όλοι οι συνάδελφοι της ομάδας μου παρόντες. Όπως είπε και ο κύριος Γκρός, έχουμε πολλές διαφωνίες μεταξύ μας. Ε, υπάρχουν συνάδελφοι όπως η και ο, η κυρία που δεν ε, συμφωνούν με την ιδέα αυτή. Και θεωρούν, όπως άλλωστε και αρκετοί στη Γερμανία, ότι η λύση που έχει ήδη δοθεί είναι αρκετά ικανοποιητική και δεν θα πρέπει να ανατραπεί τίποτα με μια συμβαστική τροπολογία. Γι' αυτό λοιπόν σας θα μπορούσε να δεχθεί ο κύριος Γκρός να κάνουμε σε τμήματα τη συμβαστική. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά προς το παρόν. E ευχαριστώ κύριο Μπράτμπορν από την ε, Συντηρητικού. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ τις δικές μου ευχαριστήσεις στον Ματιό Γκρός ε, για το έργο του και για την ε, συνεργασία, το πνεύμα συνεργασία που επέδειξε κατά την προσπάθεια επίτευξη συμβιβασμών. Όπω βλέπετε από τον αριθμό των συμβιβαστικών προτάσεων, η συζήτηση ήταν ευρύτατη ε, σε σχέση με όλη την κάμα των ε, προτινόμενων τροπολογιών. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε, κύριε Πρόεδρε, για κάθε μία από τι συμβαστικέ προτάσει για να σα πω αν η ομάδα μου είναι υπερκατά ή οτιδήποτε, θα επικεντρωθώ μόνο σε γενικά θέματα για τα οποία νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, να, επηρεάσουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Κατά βάση ε, τρία είναι τα βασικά θέματα. Είμαστε αντίθετοι πρώτον σε οποιαδήποτε πρόταση και οποιαδήποτε συμβιβαστική πρόταση που προτείνει ή θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη ρύθμιση για τις επιχειρήσεις για τον τομέα των μεταφορών, όπως και αντίθετη σε οτιδήποτε θα εξισώνεται με το να καταστεί λιγότερο ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους ανταγωνιστές της ε, από τον υπόλοιπο κόσμο. Με κάποιες συμβαστικές προτάσεις αυτό ακριβώς γίνεται. έξω και δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Δεύτερη γενική αρχή. Ήδη έχει ξεκινήσει κάπως η κατάσταση και σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές προτάσεις, κάθε τροπολογία που έχει να κάνει με την αύξηση της ε, χρηματοδότησης μας είναι, ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Δεν νομίζω θα σας εκπλήσει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ποια είναι η θέση μας. Δεν υποστηρίζουμε αύξηση σε κανέναν προπολογισμό. Είτε είναι ο προπολογισμό για τους μεταφορές, είτε για οτιδήποτε άλλο. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτό είχε ε, συμφωνήθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα για τον προπλησμό του 2012, άρα δεν μπορώ να στηρίξω κάτι που ζητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Νομίζω μια συμβιβαστική ε, μιλά για πιο ρεαλιστική χρηματοδότηση. Αυτό θα μπορούσε να εξισορροπήσει κάπως ε, τις προτεραιότητες στα πλαίσια του υφιστάμενου προπολογισμού και αυτό θα μπορούσαμε να το δεχθούμε. Εκεί που ζητείτε όμως αύξηση δεν θα στηρίξουμε τις σχετικές προτάσεις. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο και το βλέπουμε σε κάποιες συμβαστικέ προτάσεις ζητείτε δράση για τομείς που εγώ θα τους κατέτασα στον, ε, στο πλαίσιο της επικουρικότητας, δηλαδή αστικές μεταφορές ε, και συγκοινωνίες κτλ εκεί θα δυσκολευτούμε να στηρίξουμε τροπολογίες οι οποίες άμεσα ζητούν ευρωπαϊκή παρέμβαση σε θέματα τα οποία τουλάχιστον στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά από τη γνώση και σε άλλα κράτη-μέλη, είναι ζητήματα που εναπόκεινται ε, που είναι μάλλον αρμοδιότητα των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Επίσης, να πω ότι στηρίζουμε μέτρα για την περαιτέρω απελευθέρωση. Σε ό,τι αφορά τι λιμενικές υπηρεσίε, θα συμφωνήσω με την κυρία Μάισνερ. Δεν επιθυμούμε να φύγει το θέμα αυτό, αν και η αναφερμένη διατύπωση σε ό,τι αφορά την συμβαστική πρόταση κατά τμήματα, νομίζω ότι λέει θα πρέπει να διευκρινίσει η Κομισιόν τη θέση της. Αυτό δεν είναι και τόσο κακό σε σχέση με την αρχική συμβιβαστική πρόταση. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα 300 χιλιόμετρα, χαίρομαι που ο κύριος Γκρός αποφάσισε να αναφερθεί σε συγκεκριμένο νούμερο, αλλά ε, κάποιες ε, χώρες έχουν διαφορετική κατάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν ε, ένα συγκεκριμένο νούμερο, αυτό το συγκεκριμένο νούμερο που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικές, ε, διαφορετικά δίκτυα, διαφορετικές συνθήκες. Άρα ίσως να μην μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτόν τον αριθμό. Ευχαριστώ. Κράμερ για τους πρασίνους. Ja, Ήθελα καταρχάς και εγώ να ευχαριστώ θερμά τον ε, Μάτσε Γκρός και για τη διάθεση του να ε, βρεθεί μια λύση, γιατί δεν είναι πάντα δεδομένο αυτό. Βλέπω ότι προσπάθησε όχι μόνο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία για τη δική του, από τη δική του ομάδα, αλλά ώστε δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία μέσα στην Επιτροπή, ώστε να έχουμε και πιο ισχυρά επιχειρήματα ενάντια της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Οι πράσινοι φυσικά δεν συμφωνούν με όλα όσα προτείνει ο Ματιού ως συντηρητικός. Άρα θα πρέπει καθένα από την πλευρά του να τα ξανασκεφτεί και να δει πώ μπορεί να αλλάξει θέση. Ένα-δύο πράγματα στα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω το άνοιγμα από την πίσω πόρτα για τα υπερφορτηγά, για τα γιγαντοφορτηγά. Δεν μπορώ να το δεχθώ. διότι οπουδήποτε επιτρέπεται η χρήση αυτών των φορτηγών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, έχει μειωθεί κατά 50% η χρήση των συνδυασμικών μεταφορών για τα ίδια φορτία. Επομένως, σε μια περίοδο, σε μια περίοδο που πρώτο μας μέλημα είναι η κλιματική αλλαγή, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε μια τέτοια ε, εξέλιξη. Και δεύτερον, θα θέλαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τα, χρημα... για τα οικονομικά ζητήματα. Μιλάμε για επικουρικότητα, μιλούμε για κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω θα μπορούσε και να πει ότι σταματάμε να επενδύουμε στην εσφαλμένη κατεύθυνση, αλλά αλλάζουμε πορεία και επενδύουμε κατά 20% μόνο στις οδικές μεταφορές, 40% στους σιδηροδρόμους και 10-15% στις, ε, στις υποδομές για ποδήλατα, για πεζούς κτλ. Του όμως τα ποσοστά αυτά πηγαίνουν <laughs> στους ε, λιμένες περισσότερο οι επενδύσει αυτέ. Ίσως κάποιο Βέλγο ή κάποιο Ολλανδό να το αντιλαμβανόταν αυτό σε επιλογή, αλλά εγώ αδυνατό να το συλλάβω. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε τόσα πολλά ε, κονδύλια στου λιμένε, δεδομένου ότι υπάρχουν και χώρε οι οποίε δεν έχουν καν λιμένε. Και πάνω απ' όλα, γιατί θα πρέπει το θέμα αυτό να διευκρινιστεί εδώ και από αυτούς τους όρους και μόνο για τους λιμένες, όχι δηλαδή για, τους, ε, για τις λοιπές ε, μεθόδους για τα λοιπά μέσα μεταφοράς. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η αναφορά εδώ συγκεκριμένα. Επίσης, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές ε, ε, σιδηροδρομικές τροχές οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Πολωνία, Γερμανία, σε διαφορετικά ποσοστά και σε άλλες χώρες μέλη, στις οποίες θα μπορούσαμε να επενδύσουμε για να τις ε, αναζωογονήσουμε και να τις ε, ανακαινήσουμε. Φερρυπίν, το Ανόβερο, το Αμβούργο, η Βρέμη στη Γερμανία, όπως και πολλά άλλα, θα μπορούσαν ως λιμένες να συνδέονται με συνδυοδρομική γραμμή μεταξύ τους για να διευκολύνονται οι μεταφορές. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στην ιστορία των ε, λευκών βίβλων. Ε, η πρώτη υπό τον ε, Κίνοκ είχε σαν όραμα την μετάβαση του βάρους από τις οδούς στο σιδηρόδρομο. Μετά είχαμε την πρόταση για τη συλλειτουργικότητα, co-modality που δεν ξέρω ακριβώ πλέον τι σημαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, σήμαινε ταυτόχρονα και την εισαγωγή στον τρόπο με το μεταφορών των ε, ε, πλοίων, τη συντροπικότητα δηλαδή. Και στη συνέχεια αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με τα δίκτυα. Συμφωνήσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο, θυμάμαι την κυρία Γέντσεν που έλεγε δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσω εγώ με τον Γκράμερ» και όμως τελικά επέμεινε, αγωνίστηκε και κατάφερε πολλά θετικά πράγματα για, το, για τις μεταφορές και στο ε, θέμα των, ε, του προϋπολογισμού που μας έψηκαν σύμφωνος. Ξέρω βεβαίως ότι η Δανία είναι επίπεδη χώρα. Ένα σημείο λοιπόν από όλα αυτά, γιατί θα ήθελα να πω ότι γενικά είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, αλλά να υπογραμμίζω ότι έχουμε ιδιαίτερα ε, να εκπρέσουμε την ευγνωμοσύνη μας, Ματιού, για, την, ε, για τον περιορισμό της χορύπανσης, που δεν τώρα πουθενά και που όμως βλέπω ότι επανέρχεται σε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, εμφανίζεται διαρκώς. Διότι αν δεν επιληθεί το πρόβλημα αυτό της ρήπανσης, δεν θα έχει μέλλον ο σιδηρόδρομος και βεβαίως η, κλιματική, η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαιτέρως και εσένα και όλους τους συναδέλφου που συμπεριλάβατε αυτή την έννοια γιατί στην αρχή των αγώνων μας ήμασταν κάπως ε, μόνοι στο Κοινοβούλιο, μόνο εμείς οι πράσινοι επιδιώκαμε αυτό το ζήτημα της ε, μείωσης χορύπανσης. Αλλά τώρα βλέπω ότι έχει προχωρήσει πολύ. Ο κύριος Κανσιάν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Γκρός ε, για το πολύ σημαντικό του έργο. Πιστεύω ότι έκανε σημαντική δουλειά και κατάφερε με αυτήν ε, να ορίσει ένα σωστό πλαίσιο. Θα επιμείνω σε δύο παρατηρήσεις σε σχέση με την ε, συμβιβαστική 10 όπου μιλάμε για ομόλογα εκτέλεση έργων ειδικότερα για αυτό το όρο Project Bonzo, ομόλογα εκτέλεση έργων, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες που ίσως να μην έχουν μόνο μία ερμηνεία στην πρακτική ζωή και συνεπώς να οδηγούν σε παρανοήσεις. Ο φάκελος που παρουσίασε η Κομισιόν, η Επιτροπή με την ονομασία Project Bonds είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά προεριορίζεται σε ένα σύστημα διασφαλίσεων. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να κάνουμε ένα βήμα πέρα από τις διασφαλίσεις προς ε, αυτό που θα μπορούσαν να είναι τα πραγματικά ομόλογα τα οποία θα επηρεάσουν τις επιμέρους δραστηριότητες των επιμέρους έργων χρηματοδότησης που δεν καλύπτονται από την πρώτη παραχώρηση το παραπάνω βήμα είναι να ξεπεράσουμε τα 50 δις που προβλέπονται στο Connecting Europe Facility. Να πάμε πέρα από αυτό και αυτή είναι η προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουμε, διότι όλες οι δραστηριότητες υποδομής ε, δεν μπορούν να περιοριστούν στην αηφορία. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να αναφέρω αφορά τη συμβιβαστική 28 που αναφέρθηκε από τον κύριο Γκρός και από τον κύριο Ελκαλντράουι. Πιστεύω ότι εδώ χρειάζεται ομογενοποίηση ε, των όσων ψηφίσαμε πριν από λίγο καιρό για τους σιδηροδρόμους. Μαζί με τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή ε, για τις 31 2012 για την ε, Μπαν λέει το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για την απελευθέρωση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μεταφέρουμε το ίδιο πράγμα ώστε να υπάρχει ομοιογένεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Άλισον. Γιώλα Σάντερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους συνεισηγητές για την προσπάθεια που έκαναν για αυτή την ε, ατελείωτη λίστα τροπολογιών. Έχουμε εδώ μια πρόταση πιο ευανάγνωστη με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να υποδείξω δύο μικρά προβλήματα στο συμβαστική 4 προσπαθώντας να βελτιώσουμε κάποιες θέσεις παραβλέψαμε τη δική μου τροπολογία όπου πρότεινα Ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε κοινωτικό επίπεδο, αλλά και στη Γερμανία πρόσφατα με, με το Stuttgart Project πιστεύω χρειάζεται να προωθήσουμε κάτι μέσα στο κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση, κάποια ανακοίνωση, ε, στρατηγική ανακοίνωση και διαβούλευση με τους πολίτες ένα διαρθρωμένη μορφή επικοινωνίας με τους πολίτες. Αυτό θα πρέπει να προωθεί η Επιτροπή. Αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στην τροπολογία 4 και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Γκρός να το λάβει υπόψη στην τροπολογία 9 έχει συμπεριλάβει την πλευρά των logistics. Ό,τι έχει να κάνει με τα logistics, με την επιμελητία έγινε ένα φόρουμ συζήτηση για αυτό το θέμα πριν από κάποιο καιρό. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε όμως να υπάρχει κάποια συνέχεια σε αυτό, όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επιμελητία, με την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλιώ. οτιδήποτε χρειάζεται, ε, σχετίζεται με την ε, εφαρμογή μεγαλύτερης αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα προμηθειών. Θα πρέπει λοιπόν πιστεύω η τροπολογία 9 να γίνει πιο συγκεκριμένη και όχι τόσο αφηρημένη. Πιστεύω θα ήταν καλό το Κοινοβουλίο να υιοθετήσει μια πιο ομόφωνη και πιο ισχυρή θέση όσον αφορά το status διότι εάν απομακρυνθεί από αυτή την ε, θέση σημαίνει είναι σαν να είναι υπέρ των μεγάλων φορτηγών. Ε. Ο κύριος Φλέγκενσάιν. Ε, πολύ. Πρόεδρε, κύριε Μπρος, Μπρος. Ευχαριστώ πολύ για την καλή αυτή έκθεση και την πολύ καλή αυτή έκθεση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξή. Είναι πολύ σημαντική βεβαίω η μακροπρόθεσμη στόχη στον τομέα των μεταφορών, αλλά δεν επαρκούν. Γι' αυτό θα πρέπει κατά διαστήματα να επαληθεύουμε τους στόχους μας. Η ιδέα του use it or lose it, ότι μπορεί να χαθεί δηλαδή δυνατότητα αξιοποίηση ενό πλεονεκτήματο, νομίζω ότι είναι σωστή και θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Επίσης, η σχέση με τις παραμεθόριες περιοχές έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ε, ισότιμη μεταχείριση των ε, περιοχών αυτών. Ένα άλλο σημείο στο οποίο περιμένουμε πιο πολλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα, με όσα έχει μέχρι τώρα ε, πράξη θα ήταν η ιδέα της ασφάλειας με μία πιο εναρμονισμένη, με μία πιο ε, ομοιογενοποιημένη προσέγγιση, διότι τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι μόνο ένα ε, μοσαϊκό από διαφορετικές νομοθεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ για άλλη μια φορά στην, ε, στον τομέα της κοινωνικής εξασφάλισης που δεν καλύπτεται και όσο δεν υπάρχει αυτή δεν μπορώ να δεχθώ απελευθέρωση στις χερσαίες μεταφορές και επίσης μαζί με την τροπολογία 26β που ανέφερε ο κ. Ελκατράου ότι δεν θα υποστηρίξουμε γιατί συνεπάγεται επιπλέον απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών που δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα κοινωνικές διαγραφές και μετά μια λύση λογική, ορθολογική. Άρα προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προσπαθήσει να ανοίξει για τρίτη φορά ένα βαρέλι του οποίου το καπάκι θα μπορέσει εύκολα να ξανακλείσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τιτσάου. Ευχαριστώ την Προεδρία, ευχαριστώ και τον κύριο Γκρός και για την πολύ καλή του συνεργασία. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Οι τροπολογίε 1, 19 και 123 δεν βρίσκονται στη συμβιβαστική ιδίω. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία για αυτέ τι δύο τροπολογίε. Η 119 δείχνει τη διαφορά μεταξύ την ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών στις νεότερες, ε, ε, στα νεότερα κράτη-μέλη και στα παλιότερα κράτη-μέλη και η 123 δείχνει το δυναμικό, τον εκμετάλλευτο δυναμικό στην περιοχή του Δούναβη και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία διότι δεν καλύπτονται από τη συμβιβαστική 8. Ε, ευχαριστώ για την Κομισιόν η κυρία Βιέγκα. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά αξιότιμα μέλη. Εδώ μιλάμε για την έγκριση της έκθεσης ε, της Επιτροπής για την ε, πολιτική για τις μεταφορές. Συγχαίρω ε, τον εισηγητή για το έργο του και για το πώς χειριστήκε τις πάρα πολλές τροπολογίες. Η έκθεση δείχνει ότι συμμερίζεται το Κοινοβούλιο, τη μακροπροθεσμή οπτική της Κομισιόν για τις μεταφορές και σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις συμφορήσεις οι μεταφορές αποτελούν το σκελετό της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει ε, στο θεματολόγιο το 2020 και στην ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να γίνει αγωνιστικότερο στο τομέα των μεταφορών για, στο, για τις επιχειρήσεις. υποστηρίζει το Κοινοβούλιο ε, πιο αποδοτικές μεταφορές από ενεργειακή και μείωση των εκπομπών ε, καυσαερίων. Είναι πολύ σημαντική η εκθέσή σας, ε, ειδικότερα από πολιτική πτυχή. Φυσικά θέτει φιλόδοξους στόχους και ζητεί άμεσες δράσεις. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχω ξαναπεί σε σας πολλές φορές ε, για το πώς, ποια είναι η άποψή μας για τους άμεσους στόχους και τους στόχους του 2020. Φυσικά είναι δική σας απόφαση να κάνετε κάτι τέτοιο. Θα θεωρήσουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μεγάλη ενθάρρυνση εκ μέρους και ήδη έχουμε ξεκινήσει με μεγάλη χαρά. Έχουμε να σας πούμε ότι το 20% των πρωτοβουλειών έχουν ήδη εγκριθεί ή προχωρήσει αρκετά. Να σας αναφέρω για το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης ε, για τις μεταφορές, το πακέτο για τα αεροδρόμια και τις κοινέ αρχές για τα δικαιώματα των επιβατών. Κατά βάση το ευρύτερο πρόγραμμα μεταφράζεται σε πολλές προτάσεις της Κομισιόν για το έργο της για του χρόνου και κατά βάση επισημαίνουμε ότι θα γίνουν πολλά περισσότερα με το πακέτο για τους σιδηροδρόμους και την πρωτοβουλία για τα εναλλακτικά καύσιμα. Θα ήθελα επίσης να σας πω, κύριε Γκρός, ότι είμαστε υπέρ της επανεξέτασης των, αεροδρο... των υπηρεσιών αεροδρομίων και θα το βρείτε στο πρόγραμμα της Κομισιόν για το 2013. Επίσης θα πρέπει να δείτε το πρόγραμμα εργασίας που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ο κύριος Μπαρόσο. Όπως λέει η Κομισιόν στη Λευκή Βίβλο, κατά βάση το να περικόψουμε την κινητικότητα δεν αποτελεί επιλογή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω δύο παρατηρήσεις όσον αφορά την έκθεση που γνωρίζετε ήδη καλά. Θα θέλαμε μια μικρή αλλαγή στην παραγραφά 15 της έκθεσης που αφορά ε, αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών στις οδικές μεταφορές. Το κανονιστικό αυτό πλαίσιο εξυγχρονίστηκε πρόσφατα μετά από σχηνοτενή συζήτηση των συνομοθετών από το 2006. Ο τομέας τώρα ζητάει σταθερότητα και εναρμονισμένη εφαρμογή των υπερχόντων κανόνων. Συνεπώς θα σας ζητήσω εδώ να διατηρήσουμε μόνο το δεύτερο κομμάτι της παραγράφου που ζητάει εναρμονισμένη ερμηνεία της υλοποίησης και θέση σε ισχύ. Και το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω αναφέρεται στην παραγραφό 18 σε σχέση με την ε, έγκριση σιδηροδρομικών οχημάτων και όπου ζητείται να μην διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες. Στην πραγματικότητα δύο μήνες μας φαίνεται πολύ φιλόδοξο. Πιστεύουμε ότι η περίοδος έξι μηνών θα ήταν πιο ρεαλιστική και πιο αρμόζουσα. Αυτά είναι κατά βάση τα συμπεράσματά μου. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε μαζί ένα σωστό αποτέλεσμα για τις πρωτοβουλίες της Λευκής Βίβλους, για καλύτερη κινητικότητα με πιο ενεργειακά αποδοτική και ξανά συγχαρητήρια στον κύριο Γκρός και στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Για αυτή την έκθεση ευχαριστούμε. Κύριε Γκρός. Σύντομα Πρόεδρε, για μια φορά. Ευχαριστώ πολύ και για τις ε, λιμενικές υπηρεσίε, Δεν ήθελα να περάσω στα όσα είπε η Επιτροπή μόλι τώρα. Πρόγραμμα εργασία 2012 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή, το οποίο δείχνει ότι είναι διατεθειμένη υπό τι νομοθετικέ, Τι μεγάλη, τι απαστράψω ατμόσφαιρα που έχουμε σήμερα εδώ πέρα. Ε, βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει πρόταση αυτή υπό τι νομοθετικέ προτάσει. Και άρεσε ήταν σκόπιμο να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να πράξει πριν έρθει η ώρα για την κατάθεση της ε, νομοθετικής προτάσεως. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα στις ομάδες να το ξανασκεφτούν αυτό με το 26Β. Γιατί το μόνο που στάει είναι από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για το τι έχει ε, σκοπό να πράξει. Δεν νομίζω ότι θα το μετανιώσετε αν ε, δεχθείτε αυτή την πρόταση. Λοιπόν, ξανασκεφτείτε το σας παρακαλώ. Για το άλλο δεν έχω καμιά αντίρρηση. Μπορούμε να το σημειώσουμε στην, ε, στο κατάργο των ψηφοφοριών ε, εάν η κυρία Τιτσάκη, και η κυρία Γιάλα Σέντερ ζητούν μία τροπολογία που δεν θεωρούν ότι καλύπτεται από την συμβαστική τροπολογία να επανέλθει στον κατάλογο δεν έχω καμιά αντίρρηση. 160 Φερρυπίν για την κυρία Γιάλα Σέντερ. Ας ψηφιστούν αυτές οι δύο τροπολογίε. Ας μην θεωρηθεί δηλαδή ότι καλούνται από τη συμβαστική. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Αν και δεν θέλω να πω ότι ο σταθμό του Τχάρτη 21 δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα για ε, μίμηση. Και θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά για τον κύριο Κράμερ και τα ποσοστά. Στο παρελθόν είχαμε ήδη συστήσει τη στάθμιση του ε, σιδηροδρομικού δικτύου και ήδη νομίζω έχει εγγραφεί και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι ισχύει ακόμη αυτή η αναλογία, το 40% δηλαδή για τους σιδηροδρόμους. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, είναι γνωστά. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι εάν νέα σχέδια ε, εγγραφούν στα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα και αφορούν του σιδηροδρόμους, ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε μια νέα διαφορετική στάθμιση, αλλά αυτό θα συνδυαστεί και με την λυπή συζήτηση που θα πρέπει να ξεκινήσει για τα διευρωπαϊκά δίκτυα γενικότερα και τη χρηματοδότησή του βεβαίω. και επίση ενδέχεται αυτό να οδηγήσει και σε αύξηση τη αναλογία ε, που αντιστοιχεί στο σιδηρόδρομο. Όλα αυτά τα λέω προσωρινά, προς το παρόν. Γιατί θα δούμε πώ θα προχωρήσει η κατάσταση. το ποσοστό για τα ποδήλατα. Εγώ δεν έχω μια αντίληση γιατί είμαι λάτρος του ποδηλάτου, αλλά ίσως δεν θα ήταν εύκολο να ανατραπεί η συμβαστική τροπολογία στην οποία έχουμε καταλήξει. Ίσως το είμαι σε μια αιτιολογική σκέψη ή παρατήρηση να το εισάγουμε. Σαν ιδέα. Ο κύριος Κράμερ κάνει παρατήρηση που δεν ακούγεται. Για δε την Επιτροπή νομίζω ότι είναι αντιληπτό το τι λέει. Δεν θέλει να ανοίξει το θέμα της διάρκειας και του χρόνου ανάπαυσης. Διάρκειας εργασίας και χρόνου ανάπαυσης. Ε, ίσως θα ήταν καλό να επιδιωχθεί η εναρμόνιση στις, ε, στη σχετική νομοθεσία. Γιατί είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν σε διάφορες χώρες. Από την άλλη πρέπει να επισημάνω ότι όταν υπάρχουν συνάδελφοι των οποίων οι χώρες αναγνωρίζουν το δικαίωμα στον οδηγό ή την δυνατότητα για τον οδηγό να οδηγεί επί 14 μέρες συνεχώς και να επιστρέφει μόνο για ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι του, ίσως το να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό να σημάνει και ακόμη πιο μεγάλη απελευθέρωση και χαλάρωση των κανόνων για τα μέγα φορτηγά. Για να κλείσω, δεν τα υποστηρίζω. Απλώς θεωρώ ότι κράτη όπως τα ε, σκανδιναβικά φερρυπίν με τις ιδιαιτερότητες που έχουν θα μπορούσαν να διατηρήσουν την ε, δυνατότητα μέσα από την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι έχουν και τις σχετικές υποδομές, να επιλέξουν τη μία οδό ή την άλλη. Παραλαμβάνω και υπογραμμίζω ότι μπορεί να παραμείνει ζήτημα της επικουρικότητας ανάλογα με το τι προτιμάει ο καθένας, με τις συνθήκες που έχει ο καθένας. Αυτό που επιδιώκουμε εδώ δεν είναι αποδοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανοχή ζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Αύριο το πρωί ψηφοφορία. Και το επόμενο θέμα στην μέση διάταξη είναι τα δεδομένα από τους φακέλους των εμφωτών. Με την κυρία Λίχτεμπεργκερ. Νομίζω ότι έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τροπολογιών σε ε, γνωμοδότηση. 200 τροπολογίες σε γνωμοδότηση, όμως ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν έχει φτάσει. PNR λοιπόν. Και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, ε, έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ. Και αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα καυτό, ένα ζήτημα διαφιλονικούμενο, ένα ζήτημα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τον πολίτη. Πρόκειται για τα δεδομένα που προσφέρει ο κάθε ένας απλός πολίτης, προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται. Ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Όποιος σκοπεύει να ε, αναπτύξει διμερείς ε, επαφές, σας το πράξει έξω από την αίθουσα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και η συγγετριά μας προσπαθεί να μιλήσει μέσα σε όλη αυτή την οχλοβοή. Παρακαλώ. Με ησυχία όποιος θέλει να αποχωρήσει. Έλα Εύα, παρακαλώ. Λοιπόν, προσπάθησα, λέει η κυρία Λίχτενμπεργκερ, τις ε, τελευταίες αυτές εβδομάδες να συζητήσω με έτσι να που έχουν καταθέσει τροπολογίε, κάποιε λύσει που θα μπορούσαν να μας εξασφαλίσουν μείωση των τροπολογιών, πράγμα που δεν ήταν καθόλου εύκολο γιατί ήταν πολύ αποκλίνουσες μερικές φορές θέσεις. Μεταξύ του άσπρου και του μαύρου ήταν δύσκολο να βρούμε τον γκρι και να έχει και νόημα η τροπολογία συμβαστική και γι' αυτό θα ε, ήθελα να κάνω μερικά σχόλια για τις ε, τροπολογίες αυτές. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το πεδίο εφαρμογής ο σκοπός δηλαδή τον οποίο προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε και προσπαθώ ακολουθώντας και την ομολογία να περιορίσω την ε, ιδέα αυτή στην απλή, στον απλό κίνδυνο της τρομοκρατίας, μόνο εκεί θα πρέπει να γίνει η σχετική ψηφοφορία δηλαδή. Ωστόσο πολλοί συνάδελφοι δεν ήθελαν να περιορίσουν μόνο στον, ε, στην έννοια της τρομοκρατίας ή του κινδύνου της τρομοκρατίας την, ε, αυτό το πεδίο εφαρμογής. Και άρα ζητούν επιπλέον της τρομοκρατίας να συμπεριληφθεί και το ε, εμπόριο ανθρώπων, όπλων, ναρκωτικών. Αυτή λοιπόν η διαβάθμιση που προσφέρουμε, αυτή η δεύτερη λύση και Πιστεύω ότι καλύπτει πολλές από τις τροπολογίες του κυρίου Σμιτ, πιστεύω τον ικανοποιεί δηλαδή αυτή η προσαρμογή. Και έτσι σε ένα τρίτο τμήμα που πιστεύω θα καλύπτει και τις ε, προθέσεις του κυρίου Bradburn, εκεί όπου ο ίδιος αναφερόταν στα most serious crimes, και αυτό το λέω, ε, σας παρουσιάσω σε επίπεδα διαφορετικά ε, κλιμακωτά τι ε, προτάσει, γιατί θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει άλλη λύση του ή Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πεδίο, το πεδίο εφαρμογή δηλαδή. Δεύτερον, κοιτάμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καλύπτονται, ποιε πτήσει καλύπτονται δηλαδή. Μιλάμε για διεθνεί πτήσεις που έχουν απογειωθεί ή που προσγειώνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν μια πρώτη λύση. Η άλλη λύση ήταν να πούμε ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ευρωπαϊκές λύσεις, ε, πτήσεις ή ότι περιλαμβάνονται μόνο εφόσον είναι με ανταπόκριση για μια πτήση σε τρίτη χώρα. Προσπαθώ και εδώ με μια συμβαστική τροπολογία και πιστεύω θα την έχετε λάβει συνάδελφοι να καλύψω αυτές τις ε, επιλογές. Η κυρία Καμέμβερτ επίση είχε προτείνει μια, με μια προφορική τροπολογία να συζητήσουμε και για άλλα μέσα μεταφορών που δεν καλύπτονται προς το παρόν από το PNR ε, πλοία, τρένα και το καθεξής ε, να καλυφθούν. Αλλά δεν υπάρχει σχετική πρόθεση. Μια άλλη λύση συμβαστική σχετική με τη μέθοδο push and pull. Κάποιοι συνάδελφοι δηλαδή θεωρούν ότι κάθε αεροπορική εταιρεία η οποία δεν έχει τη δυνατότητα του push θα πρέπει να έχει μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο ή αλλιώς να μπορέσει να περάσει στο pull, δηλαδή να μπορεί αυτόματα να έχει πρόσβαση στα ε, δεδομένα από το σύστημα PNR εκείνος ο οποίος δεν έχει τα στοιχεία στη θέση του. Οι προτάσεις λοιπόν, ε, οι τροπολογίες Φλό, Σμιτ, Βλάστο και άλλων, Grandes, θα είχαν σαν αποτέλεσμα μια ε, συμβαστική τροπολογία η οποία αποσκοπεί κυρίως στο push, στην ιδέα του push, την οποία πιστεύω ότι ε, καλύπτουμε με το κείμενο της 2F, σίγματα Και στη συνέχεια έχουμε την εξέρεξη που επίσης συμπεριλαμβάνεται σε μια συμβεστική τροπολογία. Ένα άλλο σημείο διφλονικούμενο ήταν εάν θα έπρεπε οι αεροπορικές εταιρείε βάσει αυτής της νομοθεσίας να συλλέγουν και επιπλέον στοιχεία. Επιπλέον δηλαδή αυτών που ούτως ή άλλως καταγράφουν ε, στον κατάλογο των ε, επιβατών τους. Εδώ λοιπόν έχουμε τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων, όπου προσπαθούμε πάλι να συνοψίσουμε τις θέσεις των ενδιαφέρων συναδέλφων για να είναι πιο ξεκάθαρη ε, τα πράγματα. Η συμβαστική 6 που καλύπτει πιστεύω πολλές τροπολογίες και θα έχει και καθοριστικό χαρακτήρα για, την, ε, για, για τους αερομεταφορείς, για το τι θα πρέπει δηλαδή να πράττουν ή τι θα πρέπει επιπλέον των ιωθώτων να πράξουν. Καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να ζητούνται επιπλέον στοιχεία από όσα καταγράφονται μέχρι τώρα. Με τον Σαλφομπίρκε συζητήσαμε ιδιαίτερος το ζήτημα των κρατών μελών και τη θέση τους έναντι των κανόνων των σχετικών με το πεδίο εφαρμογή. Γιατί υπήρξε κάτι μέλη τα οποία είπαν ότι θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα και να αποκλείουν προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένα από την εγγραφή στο PNR. Έγιναν συζητήσει. Ε, πολλέ φορέ έντονες στο Συμβούλιο. Έχουμε την εντύπωση μερικέ φορέ ότι το Συμβούλιο προσπαθεί περισσότερο να καταγράψει κανόνε με ευρωπαϊκό χαρακτήρα περισσότερο γιατί δεν είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με το PNR αυτή τη στιγμή και η συμβαστική τροπολογία στην οποία προχωρούμε είναι, ε, λέει ότι εάν θέλουν να εισαγάγουν τέτοιου τύπου αποκλειστικέ διατάξει στα κράτη-μέλη, θα πρέπει αυτέ να είναι σύμφωνε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το λέμε έτσι περίπλοκα γιατί βεβαίως έχουμε να κάνουμε με την αρχή της επικουρικότητας. Ταυτόχρονα προσπαθούμε όμως να δώσουμε και αυτή τη δυνατότητα. Και στο μεγάλο κεφάλαιο του ποια είναι τα δεδομένα εκείνα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν από τα CRS. Προσπαθώ καταρχάς να βρω να διατυπώσω συμβαστικέ τροπολογίε, πράγμα που μερικέ φορέ ήταν σχεδόν και αδύνατο, γιατί είχαν μάλλον ε, συσταλτική προσέγγιση οι συνάδελφοι που αφορούσαν αυτές οι τροπολογίες. Σε ένα-δύο σημεία μόνο μπορέσαμε να κάνουμε συμβαστική, δηλαδή εκεί όπου μιλούμε για συνοδευόμενους ανηλίκους, όπου δεν μπορούν να διατεθούν όλα τα στοιχεία και έτσι έχουμε μια σταλτική ε, προσέγγιση και λέμε ότι μόνο τα άκρος απαραίτητα και διατηθέμενα ούτως ή άλλως στοιχεία μπορούν να διατίθενται, να καταχωρούνται. Και Προσπαθούμε σε ένα άλλο σημείο να δούμε και αυτό το δούμε από την ψηφοφορία, ποια είναι τα στοιχεία. Ίσως μπορέσουμε να διατυπώσουμε επαρκώς ποια είναι τα στοιχεία, τα προσωπικά, τα οποία θα καταγράφονται αποκλειστικά. Εγώ προσωπικώς προσπαθώ να είμαι στο δυνατόν πιο σαφής και σύντομη, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα αιτήματα των συναδέλφων, του οποίου και ευχαριστώ και για την καλή διάθεση και για τη συμβαστική διάθεση. Πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να έχουμε συμβαστικές τροπολογίες πιο σαφείς. Και βέβαια περιμένω να ακούσω και τα σχόλιά σας. Το κατάλογο των ψηφοφοριών δεν τον έχω ακόμη καταρτήσει. Θα προσπαθήσω στο δυνατόν πιο σύντομα και ευχαριστώ πολύ και την ε, κυρία από τη γραμματεία της Επιτροπής μας γιατί έκανε πραγματικά Ηράκλειο έργο Προσπαθώντα να, συγκεράσει, να συγκεράσει όλες αυτές τις τόσο διαφορετικές ω την προσέγγιση του τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκρός. Ε, ε, er- Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Ε, Αντικαθιστώ ένα συνάδελφο ο οποίος δυστυχώς είχε κάποιο πρόβλημα υγείας στο μάκι του και έτσι πρέπει να λάβω εγώ το λόγο του Για τις παρατηρήσεις λοιπόν της κυρίας Λίχτενμπέρκερ, το ΕΛΚ έχει να πει το εξή. Τα δεδομένα PNR δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν πολύ και να εκφραστούν με πολύ συσταλτικό τρόπο. Δεν θα συμφωνήσουμε δηλαδή να περιοριστεί υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής. Ε, αντιθέτως θα θέλαμε ένα ευρύτατο κατά το δυνατόν πεδίο εφαρμογής. Οι προτάσεις χρονικές που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε και ο κύριος Δεγκράντες, ε, ο αρμόδιος συνάδελφος, θεωρεί ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλές νομοδοτήσεις να δούμε από τις διάφορες επιτροπές και ως εκ τούτου καλό θα ήταν και πολύ πιο λογικό να μην κάνουμε τέτοιου είδου προτάσεις εμείς σε μια γνωμοδότηση. Και να αφήσουμε το θέμα αυτό στην αρμοδιότητα, στην κρίση μάλλον της καθήλυνα αρμόδιας επιτροπής η οποία είναι η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Ο κύριος Δεκράντες θεωρεί ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε πρώτο πυλώνα, αλλά με την 977 του 2008, δηλαδή τον τρίτο πυλώνα αστυνομική συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα ζήτημα νομικό περισσότερο και άρα δεν θέλω να υπησέλθω στις λεπτομέρειες για τη νομική βάση, για τις ε, ε, συμβαστικέ τροπολογίε για το σημείο, για το άρθρο 2, δηλαδή το πεδίο εφαρμογή, ε, δεν έχει αντίρρηση ο κ. Δεγκράντε ω προ τι ε, συμβαστικέ σα προτάσει. Αυτά είχα να πω εγώ εκπροσωπώντα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Χαίρετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, η κυρία Τισάου και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της. Η ομάδα των σοσιαλιστών υπέβαλε πολλές τροπολογίες. Θα θέλαμε περιορισμό του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας σε μόνο σοβαρά εγκλήματα, τα πιο σοβαρά διασυνοριακά, τα πιο σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα. Δεν υποστηρίζουμε τον ορισμό του επιβάτη ειδικότερα όταν δεν υπάρχει κάποια δίωξη κατά αυτόν, δηλαδή όταν δεν ε, είναι ύποπτη για κάτι, θα υποστήριξουμε ότι όλες οι δαπάνες που απορρέουν από αυτή την οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται από τα κράτη-μέλη. Ε, υποστηρίζουμε τη χρήση της μεθόδου pool. Όσον αφορά το διάστημα διατήρησης των δεδομένων θέλουμε μείωση αυτού του διαστήματος και πιστεύουμε ότι μια καλή συμβιβαστική λύση θα ήταν να επιλέξουμε το επίπεδο που χρησιμοποιείται στην οδηγία περί διατήρησης των δεδομένων από τους ε, φορείς ε, τηλεπικοινωνικών υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα, δηλαδή μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών. Επίσης, ε, είμαστε υπέρ του περιορισμού του τύπου των δεδομένων που, μεταδίδονται προς τρίτες, που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, Υποστηρίζουμε την κατάργηση της γραμμικής υποχρέωσης που επιβάλλεται στα κράτη-μέλη. τον έχουν μόνο 30% αντί για 60% των δεδομένων, πιστεύουμε ότι αυτή η γραμμική προσέγγιση δεν είναι εφικτή. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι στην Ολομέλεια θα χρειαστεί να υποβάλουμε μια τροπολογία λέγοντας ότι όλες οι συμφωνίες όλες οι συμφωνίες PNR που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της οδηγίας. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Λίχτεμπεργκερ, ο κύριος Δεμπάκελ για τους φιλελευθερούς. Ευχαριστώ πρόεδρε και ο κύριο Σμιτ που ήταν σκιώδης ε, για το Άλντε μου ζήτησε, δεν μπορούσε να είναι παρόν και μου ζήτησε να κάνω δύο παρατηρήσεις εκ μέρους του θα σας διαβάσω το μήνυμα που μου έστειλε το πρώτο η παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ένα πλαίσιο για εξισορρόπηση των PNR στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να οικοδομήσει τη δική του βάση δεδομένων με τις πληροφορίες επιβατών και αυτό θα ήταν μια πολύ κακή επιλογή αυτό θα ήταν η εναλλακτική λύση. Θα πρέπει να γίνουν σαφεί περιορισμοί στην ύπαρξη δεδομένων στα κράτη μελών. Αυτό αφορά τα δικαιώματα των επιβατών και τη διασφάλιση εύλογων απαιτήσεων από του αερομεταφορές. Η δεύτερη του παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ διατήρηση των απολύτω απαραίτητων στοιχείων των PNR για την επιτευχή των στόχων και των στοιχείων που ενδεχομένω θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή. Η διαβίβαση των δεδομένων κοστίζει και στους αερομεταφορείς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος περί τα δεδομένα να συμπεριλαμβάνονται στα PNR και να αποτελούν έτσι βάρος. Η τρίτη του παρατήρηση είναι ότι θέλει να ζητήσει από τα μέλη να εξετάσουν πολύ προσεκτικά το τμήμα του παραρτήματος όπου αναφέρονται τα δεδομένα PNR που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποθηκευτούν. Οι πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής των ε, υπερβαρών, ε, τα ταξιδικογραφία από όπου αγοράστηκαν τα εισιτήρια μπορεί να είναι χρήσιμε. Ωστόσο, η επιλογή θέση δεν είναι απολύτω απαραίτητη. Θα μπορούσε να διαγραφεί από το παράρτημα. Το τελευταίο σημείο που ανέφερε, που θέλει να επισημάνει, είναι ο ορισμό των τύπων εγκλημάτων για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία PNR. Επειδή είναι πολύ ευρύ το πεδίο εφαρμογή τη Κομισιόν, ελπίζει ότι η Επιτροπή Τραν θα περιορίσει το πεδίο εφαρμογή στην τρομοκρατία και σε σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα, εμπορία ανθρώπων, ε, ναρκωτικών ε, και ε, υποστηρίζει την Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λίχτεμπεργκερ και ο κύριο Μπράντμπερν. Η γνωμοδότηση αυτή μπορεί να έχει την υποστήριξή μας. Πολλοί από εμάς μπορούν να την υποστηρίξουν. Πολύ καλή γνωμοδότηση. Φυσικά υπάρχουν ένα-δυο ζητήματα που εκκρεμούν. Σε γενικές γραμμές όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε την εκθέση της κυρίας Λίχτεμπεργκ. Υπάρχουν δύο πράγματα που αναφέρθηκαν ήδη, κάποια ζητήματα που μας απασχολούν. Το πρώτο είναι το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό η κυρία Λιχτεμπέργκερ ανέφερε τρεις ε, ε, διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα πολύ σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα και μια λίστα πραγματικά εγκλημάτων που θα καλύπτονται ενδεχομένω. Ε, όποια και αν είναι η τελική μας επιλογή μέσω ψηφοφορίας, ένα πράγμα θα πρέπει να είναι σαφές δεν θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο όπω κάναμε με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα όπου υποτίθεται προσπαθούσαμε να καλύψουμε τα πιο σοβαρά εγκλήματα και τελικά ε, ε τα χρησιμοποιούσαν α πούμε για λαθρεμπορία ε, χείρων. Ε, θα πρέπει να είμαστε κάπως λογικοί ε, όσον αφορά τον περιορισμό της χρήσης αυτών των δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Το δεύτερο που έχω να πω αφορά τη μέθοδο push και pull. Ε, δεν συμφωνώ με τη χρήση της ε, μέθοδο pull. Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο push, η οποία έχει αποτελέσει και κομμάτι άλλων συμφωνιών αυτής της φύσης. Αν μη τι άλλο, για λόγους απλούστευσης, ε, η μέθοδος push είναι η ευκολότερη στην υλοποίηση. Το κύριο θέμα που μας ανησυχεί είναι ότι ορισμένες τροπολογίες αφορούν τη διαγραφή κάποιων δεδομένων θα μας απασχολούσε η περίπτωση δύο από αυτές τις περιπτώσεις οι πληροφορίες χρέωσης είναι απολύτως σημαντικό να γνωρίζουμε και οι υπηρεσίες πληροφοριών όπως γνωρίζουμε δίνουν πολύ μεγάλη σημασία για το, στον τρόπο πληρωμής ενός αεροπορικού εισιτηρίου είτε ήταν μέσω πιστοτικής κάρτας με μετρητά ή διαφορετικός ή κάποιος άλλος τρόπος. Όταν κάποιος ας πούμε αγοράζει ένα ε, εισιτήριο μιας διαδρομής με μετρητά, εκεί υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι. Αυτός λοιπόν, αυτού του είδους οι πληροφορίες δεν θέλουν να διαγραφούν. Η άλλη περίπτωση είναι οι πληροφορίες τακτικών επιβατών. Ε, θεωρώ ότι αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μπορούμε να ανοιχνεύουμε τους συχνούς προορισμούς. Θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως μέσο παρακολούθησης για την αντιτρομοκρατική δραστηριότητα. Σε γενικέ γραμμέ όμω, όπω είπα, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτή τη γνωμοδότηση και μπορούμε να υποστηρίξουμε το μεγαλύτερο κομμάτι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Σβίκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Λιχτεμπεργκέρ για το έργο της. Δεν μου κάνει έκπληξη που υπάρχουν τόσες ε, τροπολογίες ε, σε μια τέτοια γνωμοδότηση που αφορά φυσικά τη, τις ελευθερίες του ατόμου και την ασφάλεια ταυτόχρονα. Ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Είναι πολύ δύσκολο φυσικά να θέσουμε όρια. Αυτό το θέμα τη πεδίου εφαρμογή στο οποίο εργαστήκαν πολύ τα μέλη αυτή τη Επιτροπή. Όλα αυτά σχετίζονται σε μεγάλη, ε, τα, τα σοβαρά εγκλήματα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία χρησιμοποιεί την πλαστογράφηση εγγράφων, ε, την εμπορία ναρκωτικών για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της δεν μπορούμε να βάλουμε όριο μεταξύ του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Είτε λοιπόν δεν θα εφαρμόσουμε καθόλου όλο αυτό το πράγμα ή θα πρέπει να έχει επαρκές πεδίο εφαρμογή. Η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά επίσης το ζήτημα του push και pull. Με έχουν ρωτήσει πολλά πράγματα όσον αφορά τα θέματα ο κ. Μπραντβόν το είπε, είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε την τεχνική πούς γιατί είναι πιο βολική. Ωστόσο υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Από τη στιγμή που χρησιμοποιεί το push για μια εταιρεία, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία επιφορτίζεται με επιπλέον έργο, ότι υποχρεούται να κάνει περισσότερα πράγματα, και επίσης η εταιρεία καθίσταται υπεύθυνη για την πράξη με αυτόν τον τρόπο ω εκ τούτου. Εάν η εταιρεία δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσει μια τεχνική push, καθίσταται υπεύθυνη. Δηλαδή, εάν δεν εφαρμόσει την τεχνική push, σημαίνει ότι δεν έχει διαβιβάσει τα δεδομένα. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα δεν είναι δικά τη, δεν αφορούν τι δικέ τη δραστηριότητε. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια υποχρέωση για εξυπηρέτηση τρίτων. Πιστεύω ότι από νομική άποψη αυτό είναι λίγο περίεργο. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν πέρα από τη φιλοσοφική πολιτική συζήτηση για το αν θα έχουμε περισσότερες ελευθερίες ή περισσότερη ασφάλεια είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των εγκλημάτων και της τρομοκρατίας. Αλλά εδώ υπάρχουν και ζητήματα ευθύνης, ανάληψης ευθυνών που δεν έχουν αναφερθεί επαρκώς σε αυτό το έγγραφο πιστεύω. Ευχαριστώ. Κυρία Βασιλιάδα από την Κομισιόν παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στις μεμβαστικές ε, προτάσεις, ελπίζοντας να έχω μπροστά μου το σωστό κείμενο. Σε ό,τι αφορά την ατολική σκέψη 11, καλή συμβαστική, θα τη στηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά την ατολική Σκέψη 15, τη συγκεκριμένη συμβαστική πρόταση, και αυτή μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Συμβαστική για το άρθρο 2 σίγμα ταφ ή 2F λατινικό και αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε. Για το 2-1-1 τη συμβαστική είναι πολύ κρίσιμη πτυχή αυτή. Αφορά το πεδίο εφαρμογή, τον περιορισμό τη όλη πρόταση. Δυστυχώ. Ε, ε, δυστυχώς εδώ θα διαφωνήσουμε. Θα προτιμούσαμε να παραμείνει το πεδίο εφαρμογή ε, ως έχει στην πρότασή μα. Σας είχα αναφέρει στην προηγούμενη συνεδρίαση του λόγους που είναι κατά κύριο λόγο ε, επιχειρησιακοί και επειδή τα στοιχεία PNR είναι πολύ σημαντικά στην καταπολέμηση διαφόρων ειδών εγκλημάτων. Να σας θυμίσω επίσης ότι και εμείς προτείναμε να αναφέρετε serious crime και όχι all crimes, άρα περιοριζόμαστε στα σοβαρά εγκλήματα. Δυστυχώ επί τη συγκεκριμένη συμβαστική ε, προτάσεω θα πρέπει να διαφωνήσω μαζί σα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμβαστική για το άρθρο 4.3α νέα, δεν στηρίζουμε τη συμβαστική αυτή. Γιατί θα μπορούσε δυνητικά το όλο σύστημα PNR να γίνει μη επιχειρησιακό έχουμε αυτό το σύστημα για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για όλους τους ε, επιβάτες άμεσα και πρώτης άφηξης ή αναχωρησής τους. Αν τώρα ζητηθεί εξουσιοδότηση από ένα νομικό φορέα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα παρακολύσει σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία του όλου συστήματος. Το άρθρο 6 υποστηρίζουμε, για το άρθρο 15 στηρίζουμε τις συμβαστική ό,τι αφορά το παράδειγμα α σημείο 12 τη συμβαστική δεν θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε. Αυτό που λέγεται για τις γενικές ε, παρατηρήσεις. Εδώ έχουμε διάφορες ε, πληροφορίες ε, που είναι πολύ σημαντικές για την επιβολή του νόμου. Άρα εμείς προτείνουμε να παραμείνει όλο το πεδίο που αφορά τις γενικές παρατηρήσεις, ό,τι αφορά τώρα τα παραρτήμα, το παράρτημα. Είχα πει και προηγουμένως, αλλά θα το τονίσω εκ νέου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εναρμόνιση, να παραμείνει εναρμονισμένο αυτό. Είναι σημαντικό για τους μεταφορείς και στις ε, συμφωνίες που θα έχουμε με τρίτες χώρες, έχουμε ήδη ε, σχεδόν ολοκληρώσει σημεία και σε άλλες είμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης, η λίστα πρέπει να παραμείνει ίδια γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να γλιτώσουμε και χρήμα και κόπο. Μιλάω για τι αεροπορικέ εταιρείε. Σα παρακαλώ λοιπόν το παράρτημα να μην το τροποποιήσετε, να παραμείνει ως έχει. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία τιμολόγησης, όλοι ανησυχείτε για αυτά τα στοιχεία. Ακούστε, οι πληροφορίες, παραδείγματος χάρη, ο αριθμός της πιστοτικής κάρτας δεν αναφέρεται, ε, μια σειρά από χ αναφέρονται και μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία, όπως οποιαδήποτε άλλη πληρωμή που κάνετε ηλεκτρονικά. Άρα δεν είναι κάτι το τόσο κρίσιμο που θα έπρεπε να σας ανησυχεί. Έτσι λοιπόν λίγο για να το προσέξετε αυτό. Κατά τα λοιπά ευχαριστώ πολύ γιατί με τις συμβαστικές αυτές προτάσεις μας διευκολύνεται πάρα πολύ τη ζωή. Θέλεις Εύα να πεις κάτι. Ναι. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλες για τις παρατηρήσεις. Ε, να κάνω κάποια σχόλια. Γιατί δεν μίλησα για όλες τις τροπολογίες. Ήθελα να μιλήσω λίγο για την μεταβατική περίοδο. Η Κομισιόν κάνει κάποιες προτάσεις που νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο να τις ε, ακολουθήσουν οι αεροπορικές εταιρείες, να επεξεργαστούν το 30, το 60%. Ε, δεν είναι τόσο εύκολο να το μετρήσει κανείς και ούτε και πρακτικό. Δεν το θέλαμε λοιπόν. Δεύτερο σημείο η δικαστική και η αστυνομική συνεργασία. Δεν έχει αυτό να κάνει με το κανονικό καθεστώς PNR. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν παρακολουθούμε έναν ύποπτο και αν δεν λάβουμε υπόψη μας καθόλου την πρόταση αυτή, τότε μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε στο πλαίσιο της ε, δικαστικής συνεργασίας. Άρα εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να γίνει διάκριση. Τι κάνουμε εδώ. Δεν μιλάμε εδώ για δικαστική ή μάλλον για αστυνομική συνεργασία. Δεν μιλάμε για, για αστυνομική συνεργασία. Δεύτερο σημείο. Να ευχαριστήσω την κυρία Τικάο για τις παρατηρήσεις της σε σχέση με την περίοδο αποθήκευσης, διατήρησης των δεδομένων και σε ό,τι αφορά το pool και σε σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος Ερικέ, έχω τις επιφυλάξει μου. Το θέμα είναι εξετάσει βλέπω ότι κάποιοι λένε ότι το να περιμένουμε τρία χρόνια για να διορθώσει τα στοιχεία της Λουφτχάς, εντάξει δεν είναι. Θα πρέπει να το δούμε. Uh, if you have to decide between push and pull, uh, it might be a question of Αυτό το push and pull, το οθελκτικό, οστικό και ελκτικό, δεν είναι θέμα μόνο κόστους. Το θέμα είναι ποιος έχει πρόσβαση, σε ποια βάση δεδομένων και υπό ποιες προϋποθέσεις. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει τις προϋποθέσεις να τι παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά. για την κυρία Τικάου και πάλι, μακάρι να υπάρξει τροπολογία στην Ολομέλεια για την επανεξέταση όλων των διεθνών συνθήκων με βάση των συμφωνιών που θα έχουμε εμείς για το PNR. Και θα είναι ένα πολύ απαραίτητο βήμα. Τώρα για το παράρτημα. Δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να ξέρουμε το όνομα αυτού που πούλησε το εισιτήριο στον επιβάτη και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τις μεθόδους πληρωμής λοιπά. Γιατί αυτό το έχουμε ήδη ξανασυζητήσει. αν μπορούμε δυστυχώ να είμαστε σίγουροι για κάτι, είναι ότι οι τρομοκράτε ε, ξέρουν πώ να πληρώνουν για να μην μπορεί κανεί να μπει στα ίχνη του. Άρα θα σας παρακαλέσω να το εξετάσετε το όλο θέμα πάρα πολύ προσεκτικά. Απευθύνομαι τώρα στον ε, κύριο Ντεγκράντες, που βέβαια τα μηνύματά του μας τα έδωσε ο κύριος Γκρός. Αναφερθήκαμε στο παράρτημα αλλά και στα επεξεργασμένα δεδομένα. Γιατί? Γιατί αυτό επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες και Στι συζητήσει μας με τις αεροπορικέ εταιρείε, βλέπουμε ότι τι ε, ανησυχεί αυτό το θέμα και δεν είναι μόνο απλά θέμα δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και ζήτημα πολιτικής ε, του αερομεταφορέα. Πολλοί έκαναν σχετικά σχόλια. Ίσως θα έπρεπε να δουν και με την, ε, τον αερομεταφορέα στη χώρα τους, να τα συζητήσουν αυτά τα θέματα του αερομεταφορείς. Νομίζω ότι έχω κάνει ό,τι μπορούσα. Ελπίζω να έχουμε μια ξεκάθαρη λίστα ψηφοφοριών. Θα με βοηθήσουν οι συνεργάτες μου, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Και Αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ινδονησίας. εισηγητή τον υποφαινόμενο, μια από τις 19 διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν. Ε, λοιπόν, η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδονησία για ορισμένε πτυχέ των αεροπορικών υπηρεσιών που έχει ω στόχο την ευθυγράμμιση ε, τη νομοθεσία. Έχουμε ε, αυτέ λοιπόν τι συμφωνίε που προβλέπουν διατάξει που εμπίπτουν στην εθνική την ενωσιακή αρμοδιότητα Κάποια πράγματα τα έχουμε αναφέρει και στην ε, έκθεση πλαίσιο. Θέλουμε να έχουμε την ισότιμη μεταχείριση των αεροπορικών εταιριών ανεξαρτήτως της εθνικότητας του αερομεταφορέα, διατάξεις ασφαλείας επίσης, φορολογικές διατάξεις και κανόνες ανταγωνισμού. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε την διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Δεν μπορούμε να πούμε ε, παρά ναι όχι. Εγώ θα έλεγα αν κάποιος θέλει να πει όχι, να καταθέσει τη σχετική τροπολογία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Εγώ πάντως αυτό που έχω να σας προτείνω είναι να δώσουμε τη συμφωνή γνώμη μας σε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Ντεμπάκε έχει το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα. Η Γκεζίνε μου ζήτησε να σχολιάσω την συντομία να πω ότι συμφωνούμε με την έκθεση εν γέννη. Δεν έχει μείνει κάποιο θέμα ανοιχτό για εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πάντα μεγάλη χαρά με κάνω εκθέσεις. εκθέσει. Ευχαριστούμε πολύ. Εύα, πράσινα. Όλα εντάξει, κορίνα πρόβλημα. Σα ευχαριστώ. Μακάρι να είχα και στο σπίτι μου τέτοια σύμπνοια και ομοφωνία. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Ε, για τις 20 Νοεμβρίου λοιπόν, αν είχατε κάτι που να αφορά την, ε, τις μεταφορές, την Επιτροπή των Μεταφορών εν ψητής της του χρόνου, τον Ιανουάριο. Το επόμενο μας θέμα λοιπόν είναι η γνωμοδότηση της κυρίας Wills. Τροποποίηση τη οδηγία σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογία των ενεργειακών προϊόντων. άλλε, εσύ έχει τον λόγο, εσύ ανέλαβε την εκπροσώπηση. Ναι, κυρία Βίλ, πρόεδρε, μου ζήτησε να σα διαβάσω τη δήλωσή τη, γιατί έχει κάποια καθυστέρηση και δεδομένου ότι γνωρίζω τη γερμανική, σας κάνω εγώ την ανάγνωση, αγαπητά μέλη της Επιτροπής των Μεταφορών. Στη γνωμοδότησή μου για την φορολογία για, τις, ε, για τα ενεργειακά προϊόντα προτείνω την α, κύρωση αυτή τη ε, φορολογία, γιατί έχουν, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν αν θέλουν τη φορολόγηση ή όχι. Σε πρώτο βήμα, λοιπόν, δεν είναι η κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα αυτό στη φορολογία. Η διαπραγματευτική εντολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ε, σύναψη των διεθνών συμφωνιών δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαγόρευση τη φορολογία ε, για, για τα ενεργειακά προϊόντα. Ε, το 2003 λοιπόν με την ε, εκπόνηση της ισχύουσας ε, ενεργειακής οδηγίας αποφασίστηκε να αρθεί αυτή η δυνατότητα. Ο σχετισμός αλλά σχετικά στενής αναλογία ως προς τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα από τα πλοία δεν νομίζω ότι δικαιολογεί εξαίρεση από την νομοθεσία. βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, η πρόθεση μάλλον για επίλυση του προβλήματο τη φορολόγηση στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν εισαγάγει φόρο ενεργειακό στα αεροπορικά εισιτήρια. Ορισμένα λοιπόν κράτη-μέλη θα μπορούσαν να προτιμήσουν αυτή τη λύση. Μακροπρόθεσμα, εάν ε, ισότιμε συνθήκε ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων ε, μέσων μεταφορών είναι το αποσκοπούμενο, η αποσκοπούμενη λύση, μπορούμε να δώσουμε λύσεις χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές, ε, δηλαδή αυτή η πρόταση μπορεί να αποτελέσει μια προϋπόθεση για την βιωσιμότητα του συστήματος των μεταφορών. Και προσπαθώ στην ε, πρότασή μου, σε συνεργασία βέβαια με τους, με τους συντονιστές από όλες τις, ε, από όλες τις ομάδες, να κάνω και τη διάκριση μεταξύ εμπορικής και μη εμπορικής χρήσης του πετρελαίου με μια ρήτρα αναθέωση του 2015, έστω και αν αυτή δεν ήταν η αρχική μου πρόθεση. Ευχαριστώ τους και οδησίγητες για την επικοδομητική συνεργασία και ελπίζω οι συμβαστικές τροπολογίες ε, που όπου καταλήξαμε να είναι ικανοποιητικέ και να εξασφαλίσουν τη σχετική πλειοψηφία. Ω προ το κοινωτικό πλαίσιο φορολογία των ενεργειακών προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ Μάικλ. Ο κ. Κέντια για το ΕΛΚΑ. Κατάλληλη στιγμή εμφανίζεται αυτός ο φάκελος, δημιουργεί, υπάρχουν κάποια προβλήματα με δεν είναι η κατάλληλη εποχή, δεν είναι η σωστή στιγμή να προσπαθούμε να συζητάμε κάτι τέτοιο. Για να δώσω όμως μια άποψη, θα παραμείνω επικοδομητικός, έχουμε προτείνει τροπολογίες που επανεισάγουν εξαιρέσεις ε, όσον αφορά το ε, καύσιμα για επαγγελματική χρήση, όπου βρήκαμε μια συμβιβαστική λύση στον τομέα των δημόσιων τοπικών μεταφορών, ειδικότερα τα ταξί. Σύμφωνο με... Ε, πιστεύω επίσης ότι πρέπει να γίνουν εξαιρεσία τα υγρά καύσιμα. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε όσα πρότεινε η συγγήτρια, η συγγήτρια μας Βουίσσα ξεπερνάει αυτό την πρόταση της ίδιας της Επιτροπής. Αυτή είναι η δική μας άποψη και σε αυτήν θα παραμείνουμε, θα επιμείνουμε. Για τους ε, σοσιαλιστές ε, Γιάλα Σέντερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν είναι εδώ κυρία Βίλς, πάντως θέλω να την ευχαριστήσω για το έργο που έχει φέρει σε πέρασα για να συμφωνήσουμε σε αυτό το επίμαχο κείμενο που είναι γνωμοδότης Επιτροπής Μεταφορών για την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Ουσιαστικά εγγενιάζουμε, αν θέλετε τη συζήτηση, είναι όμως μια ε, συζήτηση αρκετά επίμαχη. Ε, ο κύριος Καντσιάν είπε πολύ σωστά ότι έχουμε ένα ζήτημα με το χρονοδιάγραμμα, ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε καταρχήν να είναι θετικό, γιατί θέλουμε να περιορίσουμε τον αντίκτυπο, της ε, την κατανάλωση της ενέργειας. Θέλουμε να περιορίσουμε την περιβαλλοντική ζημία. Όταν λοιπόν όλοι οι τομείς είναι σε μια δραματική κατάσταση, πραγματικά δεν μπορούμε να δίνουμε από την Ευρώπη ακόμα μια κακή είδηση. Είναι πάρα πολύ ακατάλληλη λοιπόν η χρονική στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, κυρία Βίλς και ιδίως προς εξέβρεση μιας ε, κοινής θέσης. Πρέπει να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες στις χώρες που το χρειάζονται και μέσω επίσης της ρήτρας αναθεώρησης ε, ζητούμε και από την Κομισιόν να εκπονήσει μια ειδική ναι. έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη της ε, τα προβλήματα του κλάδου. Έτσι, σε μια πιο πρόσφορη χρονική στιγμή θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν ε, την αλλαγή προς ένα πιο ακριβό καύσιμο. Σε ό,τι αφορά και τις θαλάσσιες μεταφορές, ε, εγώ πρότεινα και στο πλαίσιο αυτής της γενικής κρίσης βλέπουμε ότι θαλάσσια μεταφορά, η, μάλλον θαλάσσιες μεταφορές, οι εναέρειες μεταφορές αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες για να αντιμετωπίσουν τώρα και νέες προκλήσεις, σαν αυτές που εμείς τους επιβάλλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μα υπάρχει πρόοδος και από τον ε, Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και από τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Αν δεν υπάρξει περαιτέρω πρόοδο, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μονομερό να αναλάβει περισσότερη δράση. Αλλά επαναλαμβάνω με τα χρονοδιαγράμματα έχουμε κάποιο θέμα. Τέλο, θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά τα λιμάνια, εμεί έχουμε καταθέσει τροπολογίε με την ίδια πρόθεση, δηλαδή διευκολυνθεί η πρόσβαση στον ηλεκτρισμό στα λιμάνια. Με απλούστερο τρόπο, γιατί θέλουμε τα λιμάνια να είναι ανταγωνιστικά και να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τα σκάφτα που ελιμενίζονται σε αυτά. Νομίζω ότι συμφωνεί η κυρία Βίλσε και με κάποιε συμβιβαστικέ προτάσει πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συντάξουμε τελικά μια γνωμοδότηση που θα μπορεί να μα βρίσκει σύμφωνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σα συγχαίρω και εγώ για το εξαιρετικό πνεύμα συνεργασία ε, που διέπει αυτό το φάκελο για τους φιλελεύθερους. Είναι σημαντικό να το υπενθυμίσουμε αυτό. στόχος είναι να εξελιχθούν οι συμπεριφορές. Εδώ το ζήτημα δεν είναι να αφουσκώσουμε τους προϋπολογισμούς των κρατών. Δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτής της οδηγίας. Έχουμε εδώ ένα άρθρο για το επαγγελματικό ντίζελ. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια εύλογη μεταβατική περίοδος. Δεν μπορούμε να ζητάμε υπερβολικά πολλά. Πρέπει να είναι σαφές στο κείμενο θα χρειαστεί μια αξιολόγηση μετά από πέντε χρόνια ώστε να δούμε πότε θα ε, είναι σκόπιμο να εγκαταλείψουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ επαγγελματικού και μη επαγγελματικού diesel. Ορισμένες εξαιρέσεις έχουν προβλεφθεί εδώ. Για εμάς είναι σημαντικό να υπάρχουν υποσότιμες συνθήκες μεταξύ των διαφόρων τύπων καυσίμου. Οι εξαιρέσει λοιπόν θα πρέπει να περιοριστούν στο μέγιστο. Προβλέπουμε εδώ κάτι για τις δημόσιες μεταφορές, γιατί όχι, αλλά για τα ταξί και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες ε, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο καλή ιδέα. Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου στις εναερίες μεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές, πιστεύω πρέπει να λάβουμε υπόψη την σημερινή πραγματικότητα. Για να βρίσκεται στο προπύργιο η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ναι, να το κάνει, αλλά να, λαμβάνει, να αποφασίσει για λύσεις μόνη της, ε, αυτό θα ήταν λάθος, λαμβάνοντας ε, υπόψη τις αυτών ε, των τομέων στο πλαίσιο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα ζητώντας προσπάθειες οι οποίες δεν ζητούνται από τους ανταγωνιστές μας στις υπόλοιπες χώρες. Πιστεύουμε ότι ο ηλεκτρισμός θα πρέπει να τονωθεί όντως ε, μιλάμε γι' αυτό σε μια άλλη επιτροπή. Έχουν προβλεφθεί ε, χρονικά όρια. Είμαι και εγώ εισηγητής γι' αυτό. Χρειάζονται πολλές εξαιρέσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό το τομέα. Ε, πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα για νέες εξελίξεις και νέε μεθόδους. Ένα τελευταίο πράγμα το οποίο είχα ήδη την ευκαιρία να πω Πιστεύουμε ότι η πολιτική της Κομισιόν πρέπει να είναι ουδέτερη από τεχνολογική άποψη. Πρέπει να δώσουμε δηλαδή σε όλες τις τεχνολογίες κάποια ευκαιρία και η ανακύκλωση πρέπει να έχει τις δικές της ευκαιρίες. Πρέπει να διαφυλάξουμε την αρχή της ουδετερότητας για τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. Ε, έτσι λοιπόν προωθούμε τη συζήτηση στο φιλελεύθερη ομάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια εξέβρισης συμβιβαστικών λύσεων σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι το ECR στο σύνολό του δεν υποστηρίζει αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Συνεπώς υποστηρίζουμε την τροπολογία 11 του κυρίου Κόχο αλλά γνωρίζοντας ότι δεν θα λάβει πλειοψηφία θέλουμε να εξηγήσουμε τη θέση μας για διάφορα άλλα σημεία. Πρώτα απ' όλα ενώ θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση δεν αλλάζει οτιδήποτε ριζικά ε, στο σύστημα φορολόγησης της ενέργειας ε, και ότι μειώνει τις δυνατότητες ρύθμισης της κατάστασης ε, θεωρούμε ότι αυτή η μεταβατική περίοδος εμφανίζεται υπό πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες ε, η κατάσταση μπορεί να σταθεροποιηθεί μόνο στο απότερο μέλλον. Έτσι λοιπόν οι εξελίξεις όσον αφορούν το δίζελ και το πετρέλαιο είναι αρκετά γρήγορες, πως η βιομηχανία μπορεί να δυσκολευτεί να ε, συμβαδίσει. Όσον αφορά τι πρότασει 3, 4, 5 τη κυρία Βουίλ, όσον αφορά τι εναέρειες μεταφορέ, πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Διότι η Ευρώπη εξαρτάται επίσης και από τα ε, διεθνείς συμβάσεις ε, για τις θαλάσσιες μεταφορές και την αεροπλοεία. Δεν είναι καθόλου λογικό ε, το να σκεφτούμε ότι η αεροπλοεία μοιάζει με την αγορά των οδικών μεταφορών. επειδή το πεδίο εφαρμογής της Ευρω... Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας ε, Αεροπλοίας είναι τέτοιο που ένα αεροσκάφος μπορεί να διατρέξει την Ευρώπη χωρίς να χρειαστεί να γεμίσει με καύσιμα. Όσον αφορά την τις προτάσεις του κυρίου Ντεμπάκερς ε, για την, ουδετερότητα, την τεχνολογική ουδετερότητα, θεωρούμε ότι είναι καλές προτάσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ώστε αυτό το σχέδιο να γίνει λιγάκι πιο αποδεκτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της. Συμφωνούμε απόλυτα με την ε, έκθεση έτσι όπως προτείνεται. Τρία πράγματα έχω να πω. Το πρώτο είναι ότι το κόστος της ενέργειας αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό μοχλό για να τροποποιήσουμε τις συμπεριφορές ή να εσωτερικεύσουμε τα εξωτερικά κόστη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το ακούσαμε από τον αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας για το Περιβάλλον. Εδώ μας παρέχεται ένας μοχλός, τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Γνωρίζω επίσης καλά την κατάσταση, το τομέα των μεταφορών πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, επαγγελματίες ε, και με άλλους τρόπους ε, με το επαγγελματικό καύσιμο είναι σαν να τους λέμε ότι μπορείτε να αυξήσετε τις τιμές και εμείς θα σας δώσουμε επιδοτήσεις. Ούτως ή άλλως οι πολύ ψηλέ τιμές πετρελαίου βρίσκονται μπροστά μας. Ε, τις αναμένουμε. Οι εποχές είναι δύσκολες. Θα χρειαστεί όμως ε, να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αυτή η αύξηση είναι αναπόφευκτη. Και τέλος όσον αφορά την ενέργεια κυκλοφορία, ναι, η φορολογία της κεροζήνης είναι δυνατή σε ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκή κλίμακα. Η αλήθεια είναι όντω ότι μπορούν να διατρέξουν τα αεροσκάφη την Ευρώπη χωρίς στάση, χωρίς να κάνουν ανεφοδιασμό. δεν είναι απαραίτητο τόσο να γίνει συμφωνία σε αυτό. Θα έχουμε υποβάλει τις τροπολογίες μας που πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και που ενισχύουν κάπως ε, τη θέση της εισηγήτριας. Δεν μπορούμε να λέμε ένα πράγμα και να ζητάμε το αντίθετο. Ε, έχουμε ένα κείμενο στο οποίο πρέπει να δώσουμε κάποια γνώμη και πρέπει να δείξουμε συνοχή. Κύριε Ζήκε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω ότι είπαν οι διάφοροι συνάδελφοι. Θέλω απλά είναι μικρή λεπτομέρεια. Το σημείο με τα ταξί, επειδή είδα ότι η Κομισιόν εξαιρεί τα ταξί από τις δημόσιες μεταφορές, μου φαίνεται πολύ περίεργη αυτή η επιλογή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι να υπενθυμίσω ότι τα ταξί είναι συνήθως ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, δεν μπορούν εύκολα να αντέξουν τέτοιου είδους μέτρα. Σίγουρα πρέπει να λάβουμε μέτρα για να ενθαρρύνουμε τα ταξί προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αλλά όχι τόσο, με τόσο ισχυρές κυρώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των ταξί, ώστε να βελτιώσουμε το ενεργειακό τους προφίλ και το προφίλ εκπομπών τους αλλά δεν χρειάζεται να τα χτυπάμε διαρκώς. Έχω υποβάλει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε τον τομέα. Το εντάξει, ναι, ο κύριος... Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Και ευχαριστώ πολύ την συγκήτρια αλλά και όλους τους άλλους συναδέλφους που συνέπραξαν. Νομίζω ότι η χρήση του diesel θα πρέπει να εξεταστεί ως προς την προέλευση του μέσα από τις εξελίξεις με μια αρχή σαφή ότι όποια εξαίρεση σαχθεί δεν θα ε, διαιωνίζεται δεν θα είναι απεριόριστη. Επίσης ως προς τις ενέργειες μεταφορές. Δεν ε, με βρίσκει σύμφωνο η ιδέα που βλέπω να κυκλοφορεί και στην ομάδα μου αλλά και σε άλλες. Που την υπέρ της επικουρικότητας. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα αυτόν Και θα πρέπει να έχουμε μια πιο θαραλέα προσέγγιση. Κύριε Στεμπάκη, νομίζω ότι έχει μια καλή ε, προσέγγιση στην υπόθεση αυτή. Και κλείνοντας, θα ήθελα να στήσω μια εξαίρεση για την ηλεκτρική ενέργεια. που μπορεί να αποτελέσει μια καλή λύση και ε, για την κλιματική αλλαγή και για την καταπολέμηση της ρήπανσης. που ε, προξενούν Φερρυπίν τα πλοία που μένουν με, το, με τη μηχανή αναμένη. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την εργασία που έχει κάνει. Ε, θα ήθελα παρόλα αυτά να κάνω μια σύντομη αναφορά ε, όχι πολύ θετική για τις τροπολογίες 1 ε, και 3. Ε, η πρόταση της Επιτροπής, όπως όλοι ξέρουμε, διατηρούσε την υφιστάμενη εξαίρεση από φορολογία των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τις ναυτιλιακές μεταφορές. Όμως, οι δύο αυτές τροπολογίες θέτουν υπό αμφισβήτηση την εξαίρεση αυτή που είχε εισηγηθεί η Επιτροπή θα τοποθετηθώ ε, αντίθετα σε αυτές τις δύο. Θα ψηφίσω κατά των δύο αυτών τροπολογιών, τις 1 και 3, με την εξή λογική, κύριε Πρόεδρε. Και ποιο είναι το επιχείρημά μου. Το ενδεχόμενο να επιβληθεί φορολογία στα καύσιμα των πλοίων είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει τους πλειοκτήτες στην προμήθεια καυσίμων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν επιβάλλονται φόροι. Το γεγονός αυτό θα έχει οικονομικές συνέπειες για την κοινοτική βιομηχανία καυσίμων. Επιπροσθέτως, θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των μεταφορέων που θα συνεχίσουν να προμηθεύονται καύσιμα εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεω, αυξάνοντας έτσι τα κόστη λειτουργίας τους σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές τους, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στην επικαλούμενη μείωση εκπομπών CO2. Επιπλέον θα δημιουργηθεί έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα στην αυτιλία μικρών αποστάσεων και αντιβαίνει στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσέλκυση φορτίων από τις χερσαίες στις θαλάσσιες μεταφορές. Για αυτού του λόγου, ε, κύριε Πρόεδρε, προτίθεμαι να ψηφίσω κατά των δύο αυτών τροπολογιών, τροπολογιών 1 και 3. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κράμερ. Οι αρχέ που συμφωνούμε είναι πολύ ωραίε και καλέ. Όταν όμω έρχεται η ώρα να τι υλοποιήσουμε, εμφανίζονται όλα τα αντεπιχειρήματα. Αποφασίσαμε λοιπόν στο έγγραφο για την οδηγία του ευρώ, της Ευρωβινιέτας, την εσωτερικεύση του εξωτερικού κόστους και τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τώρα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να ε, κάνουμε αυτό το οποίο αντιστοιχεί στο 19% της φορολόγησης ε, με ΦΠΑ στα συνδρομικές μεταφορές και στις αεροπορικές μεταφορές. Μιλάμε για 30 δις είναι δυνατόν να μου πείτε λοιπόν ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε αυτό. Είναι ακριβώς η κρίση αυτή, οι δύσκολες αυτές εποχέ, εποχές, όπου ο, ο κοινός πολίτης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία και στη Γαλλία και δεχεται και η ώρα της Γερμανίας, ξέρω πάρα πολύ καλά, όπου ο κάθε πολίτης αντιμετωπίζει μια δεινή κρίση, είναι δυνατόν να ακούει να του λέμε ταξιδεύεις ίσως με το αεροπλάνο μια-δυο φορές το χρόνο αλλά είσαι εσύ εκείνος που με τη μικρή σου, την περιορισμένη συνεισφορά, την οικονομική, χρηματοδοτείς τα πλεονεκτήματα, τα προνόμια των μεγάλων, των πάρα πολύ πλουσίων για να μπορούν αυτοί δωρεάν να ταξιδεύουν, να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί λοιπόν ο φορολογούμενος, ο κοινό φορολογούμενος να πληρώνει το λογαριασμό για τους προνομιούχους εκείνους που ταξιδεύουν δεξιά και αριστερά συνέχεια και για τις δουλειές τους και για τα business τους είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο συνέχεια. Δεν θα πρέπει αυτή την αδικία να την αποκαταστήσουμε. Και επίσης, επίσης αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην ε, μείωση τη επιβάρυνση για την κλιματική αλλαγή. Άρα χρειάζεται και ισότιμη μεταχείριση, ο ισότιμος ανταγωνισμός. Εάν μου πείτε ότι το βρίσκεται πολύ δύσκολο, τότε πολύ καλά να στραφούμε προ την άλλη κατεύθυνση και να βοηθήσουμε τον κοινό πολίτη, να καταργήσουμε το ΦΠΑ και στο σιδηρόδρομο, να, να μπορούμε να τον βοηθήσουμε τουλάχιστον να το επιτρέψουμε πιο φθηνά να παίρνει το τρένο. Αυτό θα ήταν μια εναλλακτική. Αυτό θα ήταν μια, δικαιο, μια ε, δίκαιη μεταχείριση. Αυτό θα ήταν κοινωνική ε, μεταχείριση. Στο 25. Κύριε Ντεπάκερ, πολύ ωραία. Ωραία γραμμένα. Αλλά στο διατάφτα μας λέτε μόνο στις διεθνείς μεταφορές. Γιατί, γιατί, Εάν θέλουμε βεβαίω τα πάντα να γίνουν, ε, ε, μάλλον εάν ε, πρόκειται για διεθνή συμφωνία, εάν θέλουμε τα πάντα να τα εξασφαλίσουμε σε διεθνέ επίπεδο, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ. Οι Βρετανοί που μιλούν κατά τι φορολογίε, τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ, που θέλουν όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να επιβάλλουν, ακριβώ αυτό το επιχείρημα προβάλλουν. Λένε, Α, θα το κάνουμε μόνο όταν θα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί δεν πρόκειται να επιτευχθεί ποτέ παγκόσμια συμφωνία. Μα κοιτάξτε, εμεί έχουμε 500 εκατομμύρια πολίτε. οι αεροπορικέ εταιρείε που έρχονται στα δικά μα τα λιμάνια, τα ε, αεροδρόμια, συγγνώμη, παίρνουν κυροζίνη χωρί φόρο, και πάνε και έρχονται στι ΗΠΑ χωρί φόρο με κυροζήνη αφορολόγητη. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό να πούμε ότι θα το, θα το θα περιμένουμε να το ρυθμίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο τεράστιο μέγεθος στην Ευρώπη που θα πρέπει να αποδεχθεί και η αεροπορική εταιρεία η οποία θα θέλει να χρησιμοποιήσει τον αερολιμένα μας ότι θα πληρώσει και τον φόρο στην κυροζήνη όταν έρθει να γεμίσει το ρεζερβάρ του αεροπλάνου της. ο κύριο Κόχ. Έχουμε μια μεγάλη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και βλέπω ότι δυστυχώ συνεχίζουμε να συμπεριφερόμαστε όπω και στο παρελθόν. Προσπαθώ λοιπόν να δω αν υπάρχει δυνατότητα να συμβάλλουμε με νομοθετικά μέτρα ή ε, να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό λοιπόν βλέπω εγώ εδώ ότι δεν είναι απαραίτητη αυτή η φορολόγηση να, για να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης ούτε και πρόκειται να βοηθήσει γι' αυτό και θα καταψηφίσω τη σχετική πρόταση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σίμψον θέλει κανείς από την Επιτροπή να σχολιάσει. Υπάρχει εκπρόσωπος. Απλώς δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει. Θέλετε κύριε... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πράγματι ονομάζομαι Ζήφκοφ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το σημαντικότερο σημείο της συζήτησης που όπως φαίνεται είναι το γιατί η Κομισιόν δεν πρότεινε τη φορολογία της αεροπλοείας και των θαλάσσιων μεταφορών. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να το σχολιάσουμε. Θα ήθελα να πω επιπλέον ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι η οδηγία για τη φορολογήση της ενέργειας θα πρέπει να καλύπτει χρήστες και φορείς που δεν εντάσσονται στο ETS από το 2012 το σύστημα της αεροπλοείας θα συμπεριλαμβάνεται στο EU ETS. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι απαραίτητο να το συμπεριλάβουμε στην ETD. Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, πράγματι θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η σε αυτόν τον τομέα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρωτοβουλίες υπό το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η Κομισιόν προετοιμάζει μια αξιολόγηση αντικτύπου και θα έχουμε τα αποτελέσματα το τρίτο τρίμηνο του 2012 ειδικότερα αν δεν υπάρξει πρόοδο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι θα ψηφίσουμε αύριο για αυτή τη γνωμοδότηση και στη συνέχεια η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα ε, ψηφίσει 24 Ιανουαρίου. Έτσι ολοκληρώνουμε την απογευματινή μας ημερήσια διάταξη. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία των συντονιστών σε περίπου 10 με 15 λεπτά όταν θα έρθουν εδώ όλοι οι συντονιστές. Τερματίζεται εδώ λοιπόν η συζήτηση και θυμηθείτε να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας αύριο το πρωί. Ευχαριστώ.